Shall I on? Yep. Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Να σας υπενθυμίσω ότι θα ξεκινήσει η ψηφοφορία άμεσα και θα είναι ηλεκτρονική. Προεδρεύω εγώ, γιατί ο κύριος Μωραές ε, έχει ακόμα προβλήματα με τα πόδια του και βεβαίω δεν μπορεί να έρθει. Του ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση. Η κυρία Γκάλ είπε πως με χαρά θα με αφήσει να προτρέψω γιατί και εκείνη κολλείεται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ κυρία Ολμαϊρ. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ε, για τη μερική διαταξή υπάρχει αντίρρηση. Παρακαλώ κυρία μου. Με συγχωρείτε. Εμείς το ΙΕΝΕΦ e δεν θεωρούμε να μπει η Τουρκία στην ημερήσια διάταξή στη διάσκεψη των Προέδρων για την ομάδα μου την προηγούμενη εβδομάδα και είπαμε ότι δεν θα μπει στην ημερήσια διάταξη χωρίς να γίνει σωστή συζήτηση. Αυτό θέμα να γίνει είναι πολύ σημαντικό θέμα για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οπότε είμαστε κατά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Άλλες αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Να σας υπενθυμίσω συνάδελφε πως βεβαίως είναι προνόμιο του Προέδρου να καθορίσει την ημερήσια διάταξη. Αυτό το έκανε ο κύριος Μωραές και όπως ξέρετε απόψε στα... θα υπάρχει ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά και τα σχετικά θέματα τα οποία φύγει στην επιστολή του η ομάδα σας, στην επιστολή της η ομάδα σας. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν άλλες αντιρρήσεις, νομίζω η πλειοψηφία είναι υπέρ της ημερήσιας διάταξης. Σωστά σωστά και σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα. Λοιπόν, εγκρίνει τη μυρίσια διάταξη. Να πω. Δυστυχώς απόψε ε, διερμηνία στα φιλανδικά, εστονικά, λετονικά, μαλτέζικα, κροατικά και ιρλανδικά δεν υπάρχει. Αν ναι, και εγώ αναρωτιόμουν, λέω μόνο σε αυτές. Λοιπόν, με ακούτε, ναι. Σα είπα λοιπόν ποιε γλώσσε δεν έχουμε απόψε και ζητώ συγγνώμη. Αλλά όλε οι υπόλοιπε υπάρχουν. Λοιπόν. Θα ψηφίσουμε τι, τα πρακτικά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν κάποιε αντιρρήσει για τα πρακτικά τη 11 η και 12 η Απριλίου, ε, υποθέτω ότι εγκρίνονται. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Ελπίζω λοιπόν να έχετε μαζί τις κάρτες σας. Πρώτο θέμα, ορίστε. Με συγχωρείτε, άφησα την κάρτα μου στην Ολομέλεια. Θα μου τη φέρουν σε λίγο, αλλά ξεκινήστε και θα σηκώνω εγώ το χέρι. Ναι, ναι, είναι σημαντικό αυτό για την δεύτερη ψηφοφορία που είναι περίπλοκη και είναι δύσκολο αν δεν έχετε την ε, κάρτα μαζί σας. Υπάρχει χρόνος λοιπόν. Ξεκινάμε. Σχέδιο σύστασης ε, για την απόφαση του Συμβουλίου για την ε, Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Κολομβίας για απαλλαγή βίζας για σύντομη διαμονή. Η κυρία Γκαμπριέλ είναι η συγητής. Θέλετε να πείτε κάτι ή όχι. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρασε. Ευχαριστώ. 44 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Ευχαριστώ. Μετά έχουμε Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Δημοκρατίας του Παλάου για απαλλαγή από βίζα για συνομή διαμονή. Πάλι Μαρία Γκάμπριελ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 45 υπέρ, 4 κατά καμία αποχή. Σας ευχαριστώ. Και πάλι σύσταση για σύναψη συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βασίλειο της Τόγκας για απαλλαγή ε, βίζας για μικρή διαμονή άρχεται η ψηφοφορία πέρας 45 υπέρ 4 κατά καμία εποχή ευχαριστώ Λοιπόν, έλεγχος από κατοχής όπλων με εισηγητή τον Μποντίλ Βαλέρο έχουμε σχέδιο νομοδότησης η κυρία Βαλέρο θέλει να πει κάτι μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία ωραία Λοιπόν, τροπολογία 26, 27, 29, 30 και 32 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 10 υπέρ, 41 ε, κατά. Καμία αποχή απορρίπτεται. Άρθρο 1, παραγραφός 1, τροπολογία 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 18 έναντι 33. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεκτή 46 έναντι 5 οπότε περνάμε στην τροπολογία 95 υπάρχει έτοιμα για χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο αρχιτή η ψηφοφορία Α, όχι, λάθος. Πέρασε η συμβιβαστική 5. Άρα απορρίφθηκε. Λοιπόν, τροπολογία 95 σε δύο μέρη. The first falls five. It's only the second part we're voting on. Άρα ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο μέρος, τα κράτη-μέλη, θα και τα λοιπά. Λοιπόν, ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος. Α, Απορρίπτεται. Τροπολογία 101. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το έναντι. Με 50 ψήφους. Λοιπόν. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Μετά έχουμε δύο ταυτόσημες, την 103 και 104, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Οπότε η 105 καταπίπτει και περνάμε στην 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 107. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 108. Άρα ψηφίζουμε έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 109 αποσύρεται και περνάμε στην 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και γίνεται δεκτή. Μετά. Υπάρχουν δύο ταυτόσημες, η 111 και 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 113, αρχίτε η Πέρασε. Δεκτή. 115, Άρχιδη η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 116, άρχεται. Πέρας. Δεκτή με δύο ψήφους διαφορά. Εκατόν δέκα εφτά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 118. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 119. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Μέρος δεύτερο. Ε, πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο της συμβαστικής έξι, Άρχεται. Πέρας. Και το δεύτερο μέρος απορρίφθηκε. Η επόμενη λοιπόν είναι η τροπολογία 8 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 129 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 128 άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή με μία ψήφο διαφορά. 127 άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Επόμενε επόμενες είναι ταυτόσιμε. 9, 131 και 132 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Να τα επαναλάβουμε. Α, Μάλιστα. Δεν λειτουργούσε το μηχάνημα. Καλώ Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για τι 9, 131 και 132. Ψηφίστε. Ναι, τρει ταυτόσιμε είναι. Πέρας. Δεκτή. 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, δεν είχαμε κλείσει την προηγούμενη ψηφοφορία. λοιπόν, 135. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 136 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 137. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 139 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 140. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 141 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 142 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται 143 άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε δεκτή 143 α, συγγνώμη λάθος τροπολογία 10 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Άρθρο 1. Τροπολογία 144. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 145. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες τώρα. 146 και 147 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 148 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 149 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 150 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 151 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται 154. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, τώρα ψήσουμε 152, 153, 155 μαζί είναι ταυτόσιμες. Άρα έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνονται. 156. Άρχεται. Πέρας και έγινε δεκτή 158 έρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 159 έρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Εκατόν εξήντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 161. Ψήφις, άρχη η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 162 χωρίς τη ψηφοφορία. Μέρος πρώτο, Άρχη η ψηφοφορία. δεκτή και μέρος δεύτερο άρχιτη Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 άρχιτη ψηφοφορία. Α, με ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε το ΕΛΚ. Αρχίτε. Πέρας. Και απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις ε, τροπολογίες 163 και 164, ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. τροπολογία 172. 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 173. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας, Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας, Εγκρίνεται. Πάμε στην 175. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεφώς πάμε στην συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα πηγαίνουμε στην τροπολογία συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε δύο τμήματα, σε τρία μάλλον. Πρώτο τμήμα. Συμβιβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 199. Άρχεται η ψηφοφορία. Η 199. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 201. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσημες μάλλον τέσσερις ταυτόσιμες τροπολογίες, 202, 203, 204, 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη 208. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Μόλις απορρίφθηκε. Ναι. Θέλετε να ελέγξουμε. Είναι απλό. Όχι, δεν θέλω να ελέγξουμε. Η Άννα Γκόμες δεν έχει κάρτα, οπότε πρέπει να μετρήσετε τη δική της ψήφο στο αποτέλεσμα. Όταν είναι 23-23... Δεν λειτουργεί το μηχάνημά τη, μόλις τώρα το είδα. Κανονικά, αν πει στον πρόεδρο ότι δεν έχεις κάρτα, μπορούμε να το βολέψουμε. Το είπα πριν. Δεν γίνεται να πάω και εκεί για να ψηφίζω ταυτόχρονα. Συγγνώμη. Κυρία Γκόμες, θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά θα το βάλουμε στα πρακτικά, αλλά δεν αλλάζουμε την ψηφοφορία. Αυτό είναι το σωστό. Κατάλαβα όμω τι είπατε. Οπότε πάμε στη 209. Άρχεται η ψηφοφορία. 209. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 210. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 211 είναι η επόμενη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 212. Σωστά. Ναι. Ωραία. 212. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 213. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 214. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 215. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 216. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 217. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 219. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 218. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 220. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 221. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 223. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 226. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 21 και 228. Είναι ταυτόσιμες. Τις ψηφίζουμε μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πάμε στην 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 230. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 231. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 232. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ έβαλε ε, ένα νέο μέλος που δεν έπρεπε να έχει. Θα σας παρακολουθούμε. Κάντε κάτι. Έφυγαν. Ωραία. Το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Πάμε στη 233. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίας εγκρίνεται. 234. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Γι' αυτό πάμε. 251. Ναι. 251. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ταυτόσιμες τώρα τροπολογίες 252, 253, 254, 255, 256. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. Τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ταυτόσημες 257-259. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 258. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 260. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 261. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 262. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τη 263, 264 και 265 που είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε σε αλλες ταυτόσημες, ταυτόσιμες. 266-267. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Και πάλι δύο ταυτόσιμες, οι 268 και 269. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Θεολογικές σκέψεις και τα λοιπά. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες, 35 και 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 54. Ναι, είναι όλες ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Το Τροπολογία 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 58, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. απολογία 59, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβαστική 3. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τρία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. «64, 65, 66, 67 και 68 ταυτόσιμες τροπολογίες θα πρέπει να τις ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε αυτές τις πέντε τροπολογίες. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτές. 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 74. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 75. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 76. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, εγκρίνεται. υπολογείο 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 77. Ψηφίζουμε. της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 83 και 85. Ταυτόσιμες τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 87. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Αιτιολογική σκέψη 14. Το υπολογείο 88. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 89 το υπολογείο. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 90. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Και 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Ψηφίζουμε το σύνολο του νομοθετικού κειμένου όπως τοποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Συγχαρητήρια. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Uh, Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη κυρίες και κύριοι, αλλιώς θα ξενυχτήσουμε. Και έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έχει πολύ φασαρία. Κοιτάξτε, όσοι θέλετε να κάνετε κουβέντα για θέματα άσχετα με τα θέματα της Επιτροπής, βγείτε. Αν θέλετε να μετάσχετε στην σημαντική ημερήσια διάταξη που έχουμε μπροστά μας, καθίστε, μη μιλάτε και συνεχίζουμε. Προχωράμε σε κάθε περίπτωση, είτε παρακολουθείτε τι λέω είτε όχι. Επόμενο θέμα, ανταλλαγή πληροφοριών για πολίτες τρίτων χωρών και συστήματα ενημέρωσης ε, και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποινικών μητρών. Είμαι ο εισηγητή για το θέμα αυτό και το θέμα έχει να κάνει με την εξέταση των τροπολογιών. Την είχα υποβάλει σε 7 Απριλίου στην Επιτροπή. Κατατέθηκαν 41 τροπολογίε, οπότε μπορούμε να κάνουμε τώρα μια ανταλλαγή απόψεων με τον εαυτό μου καταρχά και του συναδέλφου. Θα πω δύο λόγια εγώ πρώτα και μετά θα δώσω το λόγο στου άλλου εμπειρογνώμονε. Τα σχόλιά μου θα είναι σύντομα. Πρώτον, ευχαριστώ τους άλλους σκιώδεις εισηγητές για τις τροπολογίες τους. Νομίζω, έχοντας δει τις τροπολογίες ότι θα υπάρξει συμφωνία. Δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις της σκέψης και την προσέγγιση που έχουμε. Η έκθεση είναι μια τεχνική προσαρμογή ενό υφιστάμενου συστήματος που θα βελτιώσει το εφιστάμενο σύστημα έκρης, ενώ θα συμπεριλάβει ε, θα αντιμετωπίσει μάλλον τους καταδικασμένους πολίτες των χωρών με ισότιμο τρόπο όπως ε, τους Ευρωπαίους πολίτες στα δικαστικά μας συστήματα, κάτι που παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίωνα την Ένωση. Είδα τροπολογίες για την ανάγκη χρήσης του ΕΚΡΙΣ για την ε, αναζήτηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με παιδιά. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τους πολίτες των χωρών. Επίσης, οι πληροφορίες που έχω λάβει, οι πληροφορίες των κρατών μελών που λαμβάνουν για πολίτες των χωρών που μένουν στην Ένωση θα μπορούσε να βελτιωθεί. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των πληροφοριών αυτών. Μερικέ φορέ οι, πολι... οι τρίτε χώρε εμποδίζουν τα κρατη από την περαιτέρω αποστολή των στοιχείων αυτών. Δεν ζητούμε ωστόσο το να γίνει υποχρεωτικό. Όταν ωστόσο είναι ε, δυνατό, οι πληροφορίε αυτέ θα πρέπει να διατίθενται για να παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίωνα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορώ να δεχθώ τις περισσότερες τροπολογίες του ΕΛΚ, ωστόσο δεν θέλω να υπάρξει μια κεντρική βάση δεδομένων αυτή τη στιγμή. Επίσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν σκεφτόμαστε τα ενδεχόμενα μεγάλων συγκεντρωτικών βάσεων δεδομένων ως απάντηση σε όλα τα προβλήματα ασφάλειας που έχουμε. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά ζητήματα αναλογικότητας και θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν συζητούμε θέματα ε, βάση δεδομένων. Η, το φίλτρο δι, ε, το φίλτρο, το φίλτρο αντιστοιχία μη αντιστοιχία, το hit no hit, είναι καλύτερη η λύση, κάτι που αντικατοπτρίζει και την ε, απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης για την διακράτηση μητρών δεδομένων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε περαιτέρω τι τις προτάσεις της 30 Μαΐου. Αυτή είναι η δική μου συνεισφορά κύριε και κύριοι. Οι σκιώδεις αν ε, θέλουν το λόγο, καταρχάς ο κύριος Ζάκη. Um, thank you very much, dear colleague. Ευχαριστώ συνάδελφε για την ε, σοβαρή συνεργασία που είχαμε. Από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι συμβαστικές προτάσεις που υποβάλλατε είναι εν γέννη αποδεκτές. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε ένα σοβαρό και καλό κείμενο στο εγγύς μέλλον. Υποστηρίζουμε λοιπόν εν γέννη τις συστάσεις σας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάποιοι σκιώδεις δεν είναι εδώ, δεν ξέρω αν ζήτησαν να μιλήσει κάποιος εξ ονόματός τους. Η κυρία Χέντ, επόμενη ομιλήτρια. Η κυρία Σίπελ, συγγνώμη. Με ναι, ευχαριστώ. Πρώτον, η Άννα Χέντ δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Ζητά συγγνώμη γι' αυτό και θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την ε, μέχρι τώρα καλή συνεργασία που είχαν. Βεβαίω, προς το παρόν υπάρχουν κάποια θέματα διαφωνίας μεταξύ μας. Οι σοσιαλιστές έχουν επιφυλάξει ως προς το ενδεχόμενο να προσθέσουμε τις αποφάσεις από τρίτες χώρες στο σύστημα έκρης. Για την ομάδα μας αυτό είναι θέμα ασφάλειας δικαίου. Η ανησυχία μας έγκυται στο ότι κανείς δεν θα είναι υπεύθυνο για να εξασφαλίζει ότι είναι ακριβή η πληροφόρηση αυτή και για να διορθώσει τα ανακριβή δεδομένα. Επιπλέον, δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν πληροφορίε για μη καταδικασμένα μέλη τη οικογένεια στο σύστημα έκρησης. Τέλο, θέλουμε να αποφύγουμε τη διάκριση μεταξύ πολιτών της Ένωσης που έχουν μία ηθαγένεια και πολιτών της Ένωσης που έχουν η ηθαγένεια και ενό κρατου μέλους και μια τρίτη χώρα. Για το λόγο αυτό διαγράψαμε τμήμα τη αρχική πρόταση. Άλλε πολιτικέ ομάδε έφεσαν αντίστοιχε ανησυχίε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε τη τροπολογία 50 του Γιάννα Άλμπρεχτ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιντεμβέλτ. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε όσα είπε η κυρία Σίπελ. Και αναρωτιέμαι, μιλήσατε για τις ε, τροπολογίες ε, του ΕΛΚ. Βλέπω πως έχετε δεκτεί μια ε, ίσονο σημασία τροπολογία μου στις συμβαστικές προτάσεις, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα και για τις υπόλοιπες, γιατί και για εμάς η μη διακριτική μεταχείριση των πολιτών της Ένωσης έχει μεγάλη σημασία. Η συμπερίληψη των γονέων καταδικασμένων ατόμων, όχι τόσο. Στηρίζουμε τον γενικό στόχο της πρότασης και την κατεύθυνση της έκθεσής σας, αλλά τα ζητήματα αυτά είναι σημαντικά για εμάς και θα ήθελα να ακούσω την απόψή σας. Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, εγώ νόμιζα ότι θα συνεδριάσουμε αύριο και θα ήθελα να εξοικονομήσω λίγο χρόνο. Λοιπόν, αλλά θα τα πούμε μετά. Ο κύριος Ντένις Γιόγκ είναι εδώ. Όχι. Ο Γιάννα Αλμπρέχτ. Είχε κάποιος να μεταφέρει κάποιο σχόλιο τους. Ωραία, εντάξει, θα το συζητήσουμε και αύριο, όπως είπα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε. Ε, έλεγα να μιλήσω τώρα, αλλά αφού θα υπάρξει αύριο η συνεδρίαση, θα το θέσω αύριο το θέμα. Δεν το ήξερα ότι θα υπάρχει αύριο. Okay, um, now we can go... Ωραία. Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει? Ναι, μια στιγμή. Πράγματι. Παρακαλώ. Θα... Να πω κάτι. Ε, αυτά τα οποία ήθελε να πει ο Γιάνν Φίλιπ. Κοιτάξτε, εμείς ε, θεωρούμε πως θα πρέπει να βελτιωθούν... Η τροπολογία 36 είναι για να βελτιωθούν οι συνθήκες ε, τήρησης των δεδομένων. Το 45 αφορά την ίδια κριτική μεταχείριση υπηκών και η 50 επίσης, καθώς επίσης και στην, ε, η 52 η οποία αφορά τα ποινικά μετρέω σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για σκοπούς ε, απασχόλησης. Ο Γιάνν θα ήθελε να επιμείνει στην ε, τροπολογία 36 που αφορά τον διαχωρισμό των δεδομένων σε υποχρεωτικά και μη για να υπάρξει μια εναρμόνιση αποθηκεύση των δεδομένων. Δεν είναι δίκαιο να έχουμε αυστηρότερους κανόνες αποθήκευσης για πολίτες τρίτων χωρών. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των ονομάτων των γονέων. Επίσης ανισχούμε ιδιαίτερα και τα άρθρα 4α και 4β που αφορούν διακριτική μεταχείριση ατόμων με διπλή υπηκότητα. Εάν έχει κάποιο διπλή υπηκότητα κράτου μέλου και τρίτη χώρα. θεωρείται υπήκο τρίτη χώρα. Αν είναι όμω ε, υπήκο τη Ένωση, θεωρείται απλά υπήκο τη Ένωση. Αυτό είναι απαράδεκτο για αυτού που έχουν διπλή υπηκότητα. Ευχαριστώ. Thank you very much Thank you. Um... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεδομένου του προγράμματός μας και μια που έχουμε και αύριο συνεδρίαση, εγώ δεν θα ήθελα να παρατείνω την συζήτηση γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Αν λοιπόν δεν έχετε πρόβλημα, θα μείνουμε σε αυτά απόψε και θα συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση. Εντάξει. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Σημείο 9 νομικές πτυχές ε, της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, της 20 Μαρτίου 2016. Προφανώς η δήλωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και οι συντονιστές συζήτησαν την προηγούμενη φορά πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα και αποφάσισαν να προσκαλέσουν την νομική υπηρεσία να ενημερώσει τους βουλευτές για τη νομική φύση της δήλωσης. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στην νομική υπηρεσία για να μας κάνει μια παρουσίαση και μετά ευχαριστώ να σας δώσω τον λόγο για σχόλια και ερωτήσεις. Ε, βεβαίως, όπως είπα, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο. Ο κύριος Βόρεν είναι, λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Τουρκία συμφώνησαν στις 18 Μαρτίου 2016 να εγκρίνουν μία δήλωση που είχε στόχο να εκφράσει την συμφωνία τους ως προς την ανάγκη να λάβουν συμπληρωματικά μεταδράσεις για, την, για να θέσουν τέλος στην διακίνηση μεταναστών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για να παρα, τους παρατηρούν να βρεθούν άλλες λύσεις. Το περιεχόμενο των εννέα σημείων του σχεδίου δράση πρέπει να θεωρηθεί στο πλήρες νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρο τους, ώστε να ε, μετρήσουμε τον πραγματικό νομικό τους αντίκτυπο. Προς τούτο διαπιστώνουμε ότι περιλαμβάνουν κατά βάση έναν οδικό χαρτί για την διευκόλυνση της επιτάχυνσης της υλοποίησης προϋφιστάμενων υποχρεώσεων, ενώ άλλα σημεία μπορούν να αναλυθούν ως μια δήλωση προθέσεων που εκφράζεται στα πλαίσια των ε, συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να φτάσουμε στην τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών ε, διατάξεων ή την ε, διευκόλυνση ορισμένων υποεξέλιξης συζητήσεων. Ε, θα ασχοληθώ με δύο μόνο σημεία. Το σημείο 7 για τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης και το σημείο 9 όπου η Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με την Τουρκία στα πλαίσια της βελτίωσης ε, τη ανθρωπιστικής κατασταση στο δικό της Συρίας. Αυτά τα σημεία είναι καθαρά πολιτικές δηλώσει, οπότε δεν θα υπησέλθω σε αυτά. Για τα πιο ουσιαστικά θέματα της δήλωσης αυτής, επιτρέψτε μου να κάνω μια γρήγορη επισκόπηση. Ένα, σύμφωνα με το οποίο κάθε νέοι μετανάστες ε, παρά την κατάσταση που εισέρχονται μετά από τις 20 Μαρτίου 2016 στην Ελλάδα θα, επανα, θα επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Παρατηρούμε ότι η δήλωση αυτή δεν έχει επίπτωση στο περιεχόμενο των υφιστάμενων κανόνων, δηλαδή <clears throat> την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου, την οδηγία για τις επιστροφές, ιδίως τι διατάξεις της ε, που περιγράφουν τις διαδικασίες επιστροφής και τις εγγύησεις που παρέχονται για να εξασφαλίσουν την επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών ε, που βρίσκονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επηρεάζει επίσης τις δύο συμφωνίες επανεισδοχής που υπάρχουν και που είναι εφαρμόσιμες. Η πρώτη που είχε υπογραφεί το, 2016, το Μάρτιο του 2016 μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία και από την 1η Ιανουαρίου 2016 η Συμφωνία Επανεισδοχή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για την οποία ε, συνένεσε ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την απόφαση του Συμβουλίου που, ε, που έθεσε νωρίτερα την ημερομηνία υλοποίηση τη συμφωνία αυτή όσον αφορά την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Άρα η Ελλάδα και η Τουρκία υιοθέτησαν τροποποίηση στη δική τους νομοθεσία μόνο για να προσαρμόσουν την νομοθεσία αυτή ε, σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η δήλωση εδώ δεν, έχει, δεν φαίνεται να στοχεύει στην αύξηση της επιχειρησιακής, ε, των επιχειρησιακών βαρών σε ό,τι αφορά τη δικασία επιστροφής. Τώρα, Σημείο 2 βάση του οποίου κάθε, για κάθε σύρο που επιστρέφεται στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος σύρος εγκατασταθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέμε one-to-one. -one. Αυτό το one-to-one -one αυτο το one to one ερχεται σε συνέχεια μηχανισμών που επίσης προϋπήρχαν μετεγκατάστασης που υιοθετήθηκε με απόφαση ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου του 2012 και που επανήλθε το 2015. Η απόφαση αυτή υιοθετεί, συνοδεύεται από μια δήλωση του Συμβουλίου του 23 Απριλίου 2015, προχωράω γρήγορα σε αυτά, ιδίως δε υπάρχει επιτάπητος μία απόφαση του Συμβουλίου που τροποποιεί την προγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου του 2015, του 22 δηλαδή Σεπτεμβρίου του 2015 και που υιοθετεί μέτρα προσωρινού χαρακτήρα στα πλαίσια της διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ελλάδος και της, και Ιταλίας. Απόφαση που λήφθηκε μετά από πρόταση της Επιτροπής του τοποποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2016 και που έχει στόχο την ενσωμάτωση απόφαση, προγενέστης απόφαση επιτροπής που καλείται να λάβει συμπληρωματικά μέτρα για την εξασφάλιση, την ανακατανομή πιο σωστά ορισμένων μεταναστών που ήταν από αντικείμενο παλαιότερων ε, αποφάσεων, δίνοντας 50, 54.000 θέσεις ε, στο πρόγραμμα του One to One μαζί με τις 18-20.000 που είχαν εγκριθεί νωρίτερα. Το ποσό αυτό είναι, φτάνει στις 76.000 θέσεις, θέσεις διαθέσιμες για την μετεγκατάσταση για την επανεγκατάσταση από την Συρία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομική βάση της ε, πρότασης είναι το 78.3 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου το Συμβούλιο πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο, όπως ξέρω, ασχολείται με την σχετική γνωμοδότηση. Σημείο 3 η Τουρκία θα λάβει κάθε μέτρο για να αποφύγει την, ε, το να ανοίξουν νέες δίωδοι ε, εισόδου από το έδαφος της σε γειτονικές χώρες. Και εδώ πρόκειται για μια μονομερή δέσμευση της Τουρκίας ε, που προκύπτει από το κοινό πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και που εξέφραζε μόνο την ανακοίνωση της Επιτροπής και την, στα πλαίσια της συνεργασίας με την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση αυτή η μονομερής δέσμευση της Τουρκίας δεν εισάγει κανένα νέο νομικό στοιχείο. Σημείο 4. Ενεργοποίηση ενός προγράμματος ε, υιοθέτησης των διαδικασιών εθελούσιας επιστροφής. Και εδώ υπάρχει ένα προγενέστερο πολιτικό πλαίσιο ε, μια διαδικασία ε, εθελούσιας επιστροφής που είχε προγραμματίσει η Επιτροπή έχει έναν σαφή εθελούσιο χαρακτήρα καταγράφεται σαφώς αυτό και κατά συνέπεια δεν πρόκειται για μια νομική υποχρέωση. Σημείο 5. Επιτάχυνση της ε, πιο συγκεκριμένης υλοποίησης του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Το οδικός χάρτης ήδη προβλέπει τα 72 κριτήρια αναφοράς που πρέπει να τηρηθούν για να υπαρξιάσει τι της θεωρήσεων για Τούρκους πολίτες, αλλά προς τούτο και στο σημείο αυτό η δήλωση απλώς προβλέπει μια επιτάχυνση των συζητήσεων προς την κατεύθυνση αυτής της ε, ε, απελευθέρωσης, κάτι που δεν επηρεάζει και τα κριτήρια αναφοράς που πρέπει να σέβεται η Τουρκία. Και άλλωστε η δήλωση παραπέμπει ρητά στην τελική απόφαση για το θέμα αυτό που θα πρέπει να ληφθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα σας θυμίζω ότι η Επιτροπή πρότεινε, υπέβαλε μάλλον μία πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την άρση αυτή τη υποχρεώση θεωρήσεων για τουρκου πολίτες. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγή του κανονισμού του Συμβουλίου του 2001. Η αλλαγή αυτή θα γίνει με την ε, συνήθινη νομοθετική διαδικασία. Σημείο 6 επιτάχυνση της καταβολής τριών δισεκατομμύριων ευρώ που είχαν ήδη ανατεθεί, δοθεί στην Τουρκία στα πλαίσια της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες και της επιπλέον χρησιμοποίησης άλλων τριών δις μέχρι το 2018. Διαπιστώνουμε ότι στην πραγματικότητα το μόνο νέο στοιχείο εδώ είναι η εκταμίευση των συμπληρωματικών τριών δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, η δήλωση αυτή δεν θα αποτελέσει αυτή τη νομική βάση για την ε, εκταμίευση αυτής της επιπλέον χρηματοδότησης που θα γίνει μεταξύ του προπολογισμού της Ένωσης και των κρατών μελών ο επιμερισμός του οποίου δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Σε ό,τι αφορά τον, το τμήμα του προπολογισμού της Ένωσης θα γίνει εκταμίευση βάσει των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Σημείο 8. Επιτάχυνση της διαδικασίας προσχώρησης. Ε, σημειώνουμε ότι το σημείο αυτό είναι μια πολιτική, καθαρά πολιτική δέσμευση στο πλαίσιο των ενεξελίξη διαδικασιών. Άρα, επί της ουσίας, η δήλωση αυτή πρέπει να ειδωθεί υπό το φως του προϋφιστάμενου πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας μεταφράζει τον διάλογο αυτό σε συγκεκριμένε μορφές συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου ωστόσο η δήλωση αυτή, αυτή καθεαυτή δεν παράγει κανένα καμία υποχρέωση τροποποίησης νομιμοθετικών κειμένων της Ένωσης, ούτε επιβάλλει την υιοθέτηση τέτοιων αλλαγών. Όλα τα στοιχεία που θα μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο ε, πιθανών νομοθετικών αλλαγών θα πρέπει να ακολουθήσουν την νομοθετική διαδικασία που εφαρμόζεται στα πλαίσια του δικαίου της ενώσεως. Τελειώνοντας, θέλω να προσθέσω ότι τίποτα στη συμφωνία αυτή δεν επιβάλλει να υπάρξει μια διεθνής συμφωνία σχετικά. Δεν υπάρχει ζήτημα που να υπάγεται στον τομέα των διεθνών συμφωνιών. Άρα προς τούτο όλα εξαρτώνται από το βαθμό δεσμεύσεων που είναι έτοιμες να αναλάβουν, είναι έτοιμα να αναλάβουν τα συμβαλόμενα μέρη. Μπορούν κατά επιλογή τους είτε να δεσμεύσουν την Ένωση με μια δεσμευτική η νομική πράξη, οπότε θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία διεθνούς συμφωνίας που απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες στο ιστορικό της Ένωσης, είτε θα αποφασιστεί απλώς να υπάρξει πολιτική δέσμευση μόνο με μία τρίτη χώρα και κατόπιν αυτή η πολιτική συμφωνία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Ένωσης με μια πολύ συγκεκριμένη κατ' επιλογή νομική πράξη. Από την άποψη αυτή μπορούμε να σημειώσουμε ότι η δήλωση που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή έρχεται να συμπληρώσει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Μαρτίου 2016 ε, με τις οποίες τα κράτη-μέλη όρισαν τις προτεραιότητες και την πολιτική κατεύθυνση της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, κάτι που ανταποκρίνεται ακριβώς στο δικαίωμα που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει των συνθήκων να χαράσει τις στρατηγικές γραμμές και που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετεί πολιτικές δηλώσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εν ώψη της ε, σύναψης μάλλον της υιοθέτηση από κοινών δράσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι τι θα κάνω. Κοιτάζω συνεχώς την ημερήσια διάταξη και πόσο μεγάλη είναι. Πρόκειται για μια τεχνική συζήτηση. Είναι νομικά τα ζητήματα, πολύ συγκεκριμένα και έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη που είναι πιο γενικά σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά στην Τουρκία. Θα ζητήσω λοιπόν από τους συντονιστές να είναι σύντομοι, λίγα λεπτά ο καθένας και να είναι πολύ συγκεκριμένοι ως προς τα νομικά και τεχνικά ζητήματα. Τα ερωτήματα που έχουν να τα θέσουν τώρα. Και όσοι άλλοι θέλουν να θέσουν πάλι τεχνικά και νομικά ζητήματα μπορούν να το κάνουν τώρα, όμως αν θέλουμε να πετύχουμε, να καλύψουμε όλη τη μερίσια διάταξη, πρέπει να μιλήσουμε όλοι ένα με δύο λεπτά. Ε, εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Χολμάγερ. Αν σας κατάλαβα καλά, αυτό το οποίο μας λέτε σημαίνει ότι με την ε, συμφωνία αυτή δεν έχει παραβιαστεί κάποια νομική διαδικασία, αλλά θα γίνει σεβαστή η κοινοβουλευτική διαδικασία και θα υπάρξει μια τελική απόφαση για τις όποιες πτυχές αυτής της ε, συμφωνίας. Ναι, μια πολύ ωραία σύνοψη κι άλλος ε, ε, λοιπόν δικηγόρος όπως εγώ. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε από την νομική υπηρεσία μας ξεκαθαρίζει ότι το βασικό σημείο της συζήτησης δεν είναι νομικό, αλλά έχει να κάνει με τις πολιτικές επιπτώσεις. Γιατί όταν μιλάμε για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, ένα από τα θέματα, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς ε, είχαμε για διάφορους λόγους αργή πρόοδο. Υπάρχει όμως ε, φυσικά ένα πολιτικό θέμα. Να πούμε δηλαδή όχι ότι θέλουμε απελευθέρωση των θεωρήσεων, αλλά ότι την θέλουμε πολύ γρήγορα. Άρα το θέμα είναι ιδιαίτερα πολιτικό και εξαρτάται από όλα τα θεσμικά όργανα, αν θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα και εξαρτάται και από το Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να εκπληρώσουμε τις επιταγές του Συμβουλίου να γίνει αυτό γρήγορα. Τώρα που η κατάσταση έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη μετά τις τελευταίες εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας στην Τουρκία. Άρα είναι περισσότερο πολιτικό το θέμα της συζήτησης και όχι νομικό επιβεβαιώνω ότι είναι σωστό. Όπως είπα, ζητήσαμε από τις νομικές υπηρεσίες ε, να δώσουν μια πολύ καλή νομική άποψη και ε, θα ε, συνεχίσουμε να μιλάμε για τα νομικά ζητήματα. Άρα, δεν θα αρχίσουμε τη συζήτηση μεταξύ δικηγόρων. Πάμε κατευθείαν στην κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση της λεγόμενης συμφωνίας με την Τουρκία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Όπως ξέρετε, αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευση σε ψηλότερο δυνατό επίπεδο από τους πρωθυπουργού ε, των κρατών μελών με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας και παρουσιάστηκε στους πολίτες ως μια συμφωνία. Τώρα βλέπουμε πώς η Κομισιόν και το Συμβούλιο προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ότι δεν είναι πια συμφωνία των αρχηγών ε, των κυβερνήσεων, αλλά είναι κάποιο είδους δήλωση. Γιατί, προφανώς γιατί συνειδητοποιούν ότι εάν ήταν όντως μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας σε έναν τομέα όπου έχει συναπόφαση το Κοινοβούλιο, δηλαδή την ε, μετανάστευση και τον προπολογισμό, τότε έχει υποχρέωση το Κοινοβούλιο να δεχτεί ή να απορρίψει την συμφωνία. Και ας αφήσουμε κατά μέρος ε, την ε, ηθική φύση της ε, συμφωνίας η οποία κατ' ουσίαν προχωρά σε δια της βίας, σε επαναπροώθηση των ανθρώπων αυτών σε μια χώρα η οποία επιβάλλει εδαφικούς περιορισμούς στην συνθήκη της Γενέβης και οι ένοπλες δυνάμεις οποίες αυτή τη στιγμή σκοτώνουν πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορά της με τη Συρία. Να αφήσουμε κατά μέρο και το ότι η συμφωνία είναι μάλλον αντισυνταγματική και ας πούμε ανταυτού όπως το Συμβούλιο ότι είναι μία μη δεσμευτική δήλωση και όχι πια συμφωνία. Τότε τα κράτη-μέλη μας λένε σοβαρά πως σκοπεύουν να δώσουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ στον κύριο Ερντογάν χωρίς όρους και χωρίς καμία εγγύηση ότι θα κάνει κάτι. Αυτό σημαίνει δηλαδή μη δεσμευτική δήλωση ή όπως αλλιώς το πούμε. Αν είναι δεσμευτική είμαι σίγουρη πως ε, υπάρχει μία λέξη στα νομικά. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώ ε, μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά το Συμβούλιο μετά από αυτή τη φάρσα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ένστ, παρακαλώ. Ναι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά και όποιος έχει ασχοληθεί με το θέμα γνωρίζει καλά ότι όταν έχουμε μια ε, συμφωνία με την Τουρκία κάθε φορά από νομική άποψη είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Γιατί, γιατί ε, μεγάλη μερίδα των ε, προσφύγων θα έπρεπε να έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες και άλλοι όχι. Γιατί δεν είναι όλοι Σύριοι. Ε, και αυτό ε, δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν ε, αυτό παραβιάζει τη συνθήκη της Γενέβης η οποία δεν είναι δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα αλλά με τα άτομα και τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες διαβιώνει ένας πρόσφυγας. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι και η νομική βάση πρέπει να διασφαλιστεί από την Τουρκία γενικότερα. Όσοι έχουν πάει στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσαν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία για τους συγκεκριμένους πρόσφυγες που επιστρέφουν ή που έχουν ε, παραμείνει εκεί δεν τηρούνται. Άρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία ε, για την ε, τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών συμβάσεων. Ε, αυτό είναι το γεγονός. Επίσης βλέπουμε ότι σε αυτά τα θέματα εμείς τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Δεν θέλουμε την υποστήριξη του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Θέλουμε μια ξεκάθαρη δήλωση από την νομική υπηρεσία ότι θα υπάρξει μια εμπειρογνωμοσύνη και στην Ισπανία και στη Γερμανία, κάτι που στην Γερμανία αυτή τη στιγμή ε, δεν δηλώνεται ξεκάθαρα, που λέει ε, ότι αυτή η συμφωνία είναι αντισυνταγματική για την Γερμανία, αντίστοιχα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη, δεν είναι εδώ. Θέλει η κυρία Κέλλερ να μιλήσει εκ μέρους της. Ευχαριστώ. Είναι μια πολιτική συζήτηση αυτή η οποία πρέπει να γίνει, αλλά υπάρχουν και κάποιες νομικές πτυχές. Γιατί από ό,τι κατάλαβα εσείς ε, είπατε ότι δεν είναι δεσμευτικό για καμία πλευρά. Εντάξει, καλό αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα νομικά ζητήματα. Δηλαδή, τι δυνατότητες έχουμε εμείς ως Κοινοβούλιο να παρέμβουμε. Τι αρμοδιότητες έχουμε για να σταματήσουμε αυτή τη συμφωνία, δήλωση, όπως το πει κανείς. Επίσης, ε, ποιο είναι το δικαίωμά μας που έχουμε, δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί βεβαίως αυτό έχει πολλές συνέπειες για πολλούς ανθρώπους. Και το θέμα είναι μετά τι είναι, αν είναι συμφωνία, δήλωση κτλ. Αν είπατε ότι δεν είναι θεσμευτική, είναι θετικό αυτό. Επίσης, το εάν η συμφωνία αυτή σέβεται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Οδηγίας περί ασύλου και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Και νομίζω πρέπει να απαντήσουν και αυτά. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, κυρία θα ήθελα να μιλήσει για το ECR αντί Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, το ECR θεωρεί πω η συνεργασία με την Τουρκία είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να ανακουφθούν πιέσει τη μεταναστευτικής κρίση. Όμως, θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει συνεργασία με ναι, πολλές ε, τρίτες χώρες, όχι μόνο την Τουρκία. Αυτό αφορά την άμεση επαναγκατάσταση, την καταπολέμηση των τράφικερ, την ε, επανεισδοχή και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το ECR θεωρεί πως η συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να αποτελέσει μαγική λύση για όλα μας τα προβλήματα στον τομέα αυτών. Επίσης, ε, εμεί θα θέλαμε τα λεφτά που πάνε στην Τουρκία να σχετίζονται με αποτελέσματα με ξεκάθαρα μετρήσιμα μετρήσιμους όρους όσον αφορά τις επιστροφές αλλά και, τις, και αποτελέσματα στο μέτρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, έχουμε ανησυχίες για τις αυξανόμενες και συνεχιζόμενες πιέσεις στις μεσογειακές χώρες και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η έκθεση της Κομισιόν λέει πως από όταν ετέθη ενισχύ η συμφωνία είχαμε 386 επιστροφές από τα νησιά της Ελλάδος στην Τουρκία. Θεωρείτε πως πραγματικά αξίζει για τα λεφτά που δίνουμε, πως θα ήταν καλύτερα τα λεφτά αυτά να τα διαθέσουμε για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα εντός της Ένωσης, όπως ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, καλύτερες εγκαταστάσεις κράτησης, περισσότερα μηχανήματα δακτυλοσκόπησης, περισσότερα λεφτά για την ένταξη ή περισσότερα χρήματα για τις επιστροφές σε περισσότερες τρίτες χώρες. Και έχω άλλη μια ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω. Είχαμε 386 επιστροφές. Είναι ακριβές αυτό το νούμερο τόσοι άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα. Είχα την εντύπωση ότι έφτασαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο αριθμός των επιστροφών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί από δύο οπτικές τεχνικά νομικά αφενός και πολιτικά αφετέρου. Ως προς την πρώτη διάσταση νομίζω ότι υπήρξε μεγάλη σύγχυση μεταξύ του τύπου και του περιεχομένου, της ουσίας της συμφωνίας. Και απόψε αναφέρθηκε ότι η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική, ότι έχει τιμωθεί μια συμφωνία μεταξύ κρατών μελών και Τουρκία, και άρα δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί η, η κανονική διαδικασία διαβούλευση του Κοινοβουλίου. Ωραία, αν δείτε όμως το περιεχόμενο, την ουσία της συμφωνίας αυτής μεταξύ <clears throat> κρατών μελών και Τουρκίας, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ε, διεθνούς συμφωνίας, αμοιβέ ε, δεσμεύσεις σαφείς μεταξύ Ένωσης Τουρκίας. Καταρχάς το one-to-one -one. to one προβλεπει η επιτάχυνση της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Υπάρχουν δηλαδή σαφείς δεσμεύσεις και ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τον προπολογισμό της Ένωσης. Δεν μπορεί να μην είναι δεσμευτικό αυτό. Είναι κάτι που περιέχει σαφείς επιπτώσεις από μια τεχνική νομική οπτική γωνία. Γι' αυτό, αν θέλει κανείς να ε, σκεφτεί ε, κακά, το κα ύπουλα, είναι, θα μπορούσε να πει ότι το έκαναν ακριβώς για να αποφύγουν το κοινοβούλιο. Αν θέλουμε το, το θέμα να το δούμε πολιτικά, είναι σοβαρότερο το θέμα. Δεν είναι δυνατόν θεσμοί της Ένωσης να δουν τελείως από, ε, ξεχωριστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί τα κρατημέλη να κάνουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να ακούσουν την άποψή μας πριν λάβουν αποφάση, διότι αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις ό,τι αφορά την, με τις μεταναστευτικές ώρες. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορεί το Κοινοβούλιο να λάβει θέση. Ας μας πει το, η νομική υπηρεσία πώς μπορεί να παρέμβει το Κοινοβούλιο σε μια συμφωνία που έχει υπογραφεί και ήδη αποδίδει καρπούς, υλοποιείται δηλαδή. Ευχαριστώ. Κύριε Μάγερ. Λείπει. Έχουμε άλλους ομιλητές θέλω το θέμα να το συζητήσουμε εκτενέστερα με τη συμβολή της Επιτροπής. Δεν μπορούμε να φάμε όλο το χρόνο συζητώντας μόνο την ε, συμφωνία. Θα είμαι σκληρός. Θα δώσω και τον, επιπλέον, τον λόγο στους επιπλέον ομιλητές, όλοι οι άλλοι κρατηθείτε. Για να μπορέσουν να απαντήσουν και οι νομικοί μας μετά, η κυρία Γκόμες. Είναι σαφές λοιπόν πως δεν είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, είναι μια επέσχυντη, ανήθικη και παράνομη πολιτική συνεννόηση, τίποτα περισσότερο. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επεσήμανε ήδη η κυρία Βίξτρομ, αχνόηθηκε εντελώ από το Συμβούλιο για ένα ζήτημα μεγάλης ε, σημασίας καθώς έχουμε επιπτώσεις ε, και στον τομέα του υπερπολογισμού και της μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να μου πει η νομική υπηρεσία είναι το ότι ό,τι και αν είναι αυτό το πράγμα αν ε, σέβεται τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών και της Ένωσης σε ό,τι αφορά δηλαδή την σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες γιατί προφανώς παραβιάζει κάθε τέτοια υποχρέωση και οπωσδήποτε τα κράτη-μέλη είναι υπόλογα όχι μόνο η Ελλάδα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα ήδη με την εφαρμογή αυτού του πράγματος δηλαδή τις επιστροφές ανθρώπων που δεν είχαν καν την ευκαιρία να εξεταστεί η υπόθεσή τους ναι ναι ναι ναι άνθρωποι επιστράφησαν ήδη στην Τουρκία χωρίς να έχουν την ε, ευκαιρία να τους ακούσει η πατερμοστία του για τους πρόσφυγες άνθρωποι οι οποίοι κρατούνται και τους έχω δει τους έχω δει τους έχω δει κρατούνται παρανόμως και άνθρωποι οι οποίοι πυροβολήθηκαν επειδή εξεγέρθηκαν κράτη-μέλη, όχι μόνο η Ελλάδα, ε, είναι υπόλογα και πρέπει να λογοδοτήσουν ε, για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Για να μην αναφέρω την εσχρή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα πω πως βεβαίως αναφέρθηκε η συνεργασία με την Τουρκία, αλλά η Τουρκία θα έπρεπε να ε, είναι εταίρος σοβαρός. Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει και από ό,τι φαίνεται τώρα μπαίνουμε στην πολιτική ουσία της υπόθεσης, αλλά θα δούμε ε, ότι η Τουρκία ποτέ δεν είχε την πρόθεση ε, να τηρήσει τις όποιες δεσμεύσεις. Σας ευχαριστώ. Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος. Ο κύριος Χριστοφόρου. Κύριε... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία, είτε και από νομική πλευρά, είτε και από πολιτική. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε τις αλήθειες. Η Τουρκία δεν σεβάστηκε τις συμφωνίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 πήρε εισιτήριο για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ενταξιακή τη πορεία με δέσμευση να εφαρμόσει το πρωτόκολλο τη Άγκυρα. Ενώ πήρε αυτό που ήθελε, μέχρι σήμερα εδώ και 11 χρόνια δεν εφαρμόζει τη συμφωνία που υπόγραψε. Η συμφωνία επανεισδοχή. Και εδώ είναι και οι ευθύνε τη Κομισιόν και των άλλων οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ υπεγράφει η συμφωνία τη επανεισδοχή, η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία έναντι χώρα μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι τη Κύπρου. Πώ είναι δυνατόν να είναι σε ισχύ μια συμφωνία που εφαρμόζεται à από την Τουρκία και μάλιστα αφήνεται ατιμωρητή Τουρκία να προχωρεί. Πώ μπορούμε να εμπιστευτούμε την Τουρκία ότι και αυτά τα 72 κριτήρια που τάχατε θα υλοποιήσει. Ότι δεν θα είναι μόνο στο χαρτί και τελικά εκεί που θα έρθει η ώρα που πρέπει να υλοποιήσει τα κριτήρια, στην πράξη δεν πρόκειται να τα υλοποιήσει. Δυστυχώ έχουμε μια αναξιόπιστη στρατηγική εκ μέρου τη Τουρκία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να γνωρίζω πώ αντιδρά και το Ευρωκοινοβούλιο μπροστά στην προκλητική στάση τη σημερινή Τουρκία του Ερτογά που πέραν από το ότι προσβάλλει το Ευρωκοινοβούλιο στέλνοντα την έκθεση πρόοδου πίσω, προκαλεί και όλα λέγοντα ότι η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία τη και η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ούτε τη συμφωνία επανεισδοχή, αλλά ούτε και τα υπόλοιπα από τα πέντε κριτήρια τα οποία αναπομένουν το να στέλνετε το μήνυμα από την Κομισιόν ή από άλλους ότι θα γίνει συμφωνία γιατί θέλουμε να εξυπηρετήσουμε το προσφυγό που θέλουμε να το εξυπηρετήσουμε, πιστεύω είναι λαθασμένο. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία μπορεί να βοηθά τώρα στο προσφυγό, αλλά και η Τουρκία παίρνει τεράστια ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ενταξιακή της πορεία. Δεν βλάπτεται μόνο η Τουρκία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Τουρκία θετήσει τι συμφωνίε, βλάπτεται πρωτίστω και η Τουρκία και πρέπει να πάρει το μήνυμα ότι δεν δικαιούται να αθετεί τι συμφωνίε, να προσβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητά και τα ρέστα από πάνω η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, αλλά είπα ότι αυτά έχουν να κάνουν με νομικά ζητήματα και όχι πολιτική συζήτηση. Όποια και αν είναι τα αισθήματά μας, ε, αν έχουμε χρόνο θα τα δηλώσουμε, αν δεν έχουμε, καλό θα είναι να μην το κάνουμε, διότι θα μιλήσουμε με την Κομισιόν για πιο ευρεία ζητήματα που είναι πολύ πιο σημαντικά. Οπότε, ζητώ συγγνώμη όσοι θέλουν τώρα να μιλήσουν, ε, να ε, σταματήσουμε εδώ, γιατί θέλουμε να παραμείνουμε στο νομικό πλαίσιο, όπως είπα. Νομικά ζητήματα. Η κυρία Ίντεμπελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας την νομική υπηρεσία έχουν εντύπωση ότι αν ε, κοιτάξει κανεί αυτή τη συμφωνία, δήλωση, άρθρο-άρθρο, πως ε, όλα είναι καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι πως ε, δεν παρουσιαστηκε άρθρο προς άρθρο, αλλά ως ένα πακέτο. Και έχει σημασία και νομικά μιλώντα ότι η Κομισιόν μέχρι τι 19 Απριλίου χρησιμοποιούσε τον όρο συμφωνία και μετά ξαφνικά, χωρίς καμία εξήγηση, άρχισε να μιλάει για δήλωση. Η Κομισιόν λοιπόν συνειδητοποίησε απολύτως τις νομικές συνέπειες του όρου. Και είναι ανησυχητικό το ότι ε, το πακέτο αυτό ή ότι είναι τέλος πάντων περιέχει στοιχεία τα οποία από μόνο τους προϋπήρχαν ε, είναι μέσα τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν με την τακτική νομοθετική διαδικασία και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου κτλ. κτλ. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε χαρτογράφητα νερά, νομικά μιλώντας, γιατί τα κρατημέλη, κομισιόν, δεν ξέρω ποιος τελικά ε, συνυπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Το πράγμα. υπερβαίνει όλες τις ε, δομές είναι εκτός ε, κάθε δομής που έχουμε για τέτοιες ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και θεωρώ πως εντάξει, πρέπει να κάνουμε συμφωνίες με γειτονικέ χώρες και άλλες χώρες αλλά εδώ πέρα μπαίνουμε φτάνουμε στο σημείο στο οποίο τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν κάνουν ό,τι τύχει. Και δεν υπάρχει δημοκρατική εποπτεία ούτε από τα εθνικά κοινοβούλια, ούτε από τα δικαστήρια. Είναι κάτι το νεφελώδες. Δεν είμαι σίγουροι ότι αν το δει κανεί ε, άρθρο-άρθρο, οπωσδήποτε θα καταλήξει στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η νομική υπηρεσία. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω από την νομική υπηρεσία, αν δεν το δούμε άρθρο προ άρθρο, αλλά ω ένα πακέτο που το παρουσίασαν ω συμφωνία, ακόμα και αν ήταν ε, απλά κωδικοποίηση διαφόρων πραγμάτων και μετά το λένε δήλωση. Εδώ πέρα υπάρχει ένα νομικό προηγούμενο το οποίο με κάνει να ανησυχώ. Ευχαριστώ, κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση, κάποιες ερωτήσεις προς τη νομική υπηρεσία. Αξιολογήθηκαν, συγκρίθηκαν κατά στην κρίση σας οι πολλές απόψεις αυτών που θεωρούν αμφιλεγόμενοι νομικά την συμφωνία, κρίνοντας από κοινού ταυτόχρονα και τη συμφωνία και τις συμφωνίες επανεισδοχής με την Ελλάδα, αλλά και την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής. Λήφθηκε αυτό υπόψη. Τα πιο αφιλεγόμενα σημεία των νομικών όχι τυχαίων, επιφανών νομικών και οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, το UNHCR. Τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία έχουν τύχη από τη δήλωσή σας περιγραφής ως πολιτικές δράσεις και είναι τα θέματα που αφορούν το σημείο 1 ιδίως όπου συστήνεται μαζικός την επαναπατρισμός, όλοι επιστρέφονται στην Τουρκία. Τούτο δεν έχει επιπτώσει στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς δεν έχει οδηγίες. Είναι μια φράση που περιγράφει σαφώς μια δυνατότητα ομαδικής επαναπρόθεσης. Δεύτερον, διεθνής συνθήκη. Πρώτα το είπαν statement, μετά deal, μετά agreement τι, μια, μια τυχαίες λέξεις είναι αυτές. Δεν είναι δήλωση. Όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κρατών είναι διεθνή συμφωνία. Και δεν το λέω εγώ αυτό που δεν είμαι δικαστήνα. Το λένε νομομαθείς του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Μία διεθνή συνθήκη απαιτεί δημοκρατικό έλεγχο που δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση και ευρωπαϊκό έλεγχο και εθνικό έλεγχο. Και τα κράτη-μέλη μέσω των κοινοβουλίων τους πρέπει να μου ρωτήσουν σχετικά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ποιος. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω τεχνικές Ερωτήσει προ την νομική υπηρεσία. Κοιτώντα την αξιολόγηση και τα στοιχεία της αξιολογήση θέλω να αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Ενδεικτικά. Βεβαίω μπορούσα να αναφέρω κατάλογο ολόκληρο. Αλλά θα αναφερθώ σε λίγα μόνο. Παραδείγματο χάρη. είναι υπαριθμών 15. Να διασφαλιστεί επαρκής συνεργασία με τα γειτονικά κράτη-μέλη τη Ένωση με στόχο ιδιαίτερα την ενίσχυση της διαχείρισης ε, των συνόρων με τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ούτε λέξη για ένα κράτος μέλος κοντά στην Τουρκία, που συνορεύει με την Τουρκία, που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Μαυρίδη, με συγχωρείτε. Ε, εσείς μιλάτε για την απελευθέρωση της βίζας που είναι το επόμενο θέμα και θα φτάσουμε εκεί. Μήπως να το θέσετε τότε. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένα για το τωρινό θέμα, συνεχίστε. Αλλά συζητάμε άλλο θέμα. Θα μου δώσετε τον λόγο μετά, αν έχουμε χρόνο. Μάλιστα. Αλλά αν συνεχίσετε με αυτόν τον κατάλογο, δεν θα έχουμε χρόνο. Ωραία, άλλη μία ερώτηση λοιπόν. Μπορούμε, υπάρχει νομική βάση για συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης χώρας όταν αυτή η τρίτη χώρα, όταν μιλάμε για συνεργασία νομικών, δικαστικών συστημάτων, δεν αναγνωρίζει τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ε, ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Λεμπρέτον. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει καθόλου καλά και η σημερινή συζήτηση στην ουσία μας αποκαλύπτει μέσω της Τουρκίας την κρίση. Αυτό που λέγεται σήμερα μας εκπλήσει ότι δεν μπορεί να, είναι μπορεί να μην είναι δεσμευτική η συμφωνία με την Τουρκία και ότι υπάρχουν νομικά στοιχεία τα οποία έχουν ως στόχο να απαραγωνίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, Συμπεράνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή απλώς παραβιάζουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι Προσπαθούμε να σώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία η οποία παραβιάζει το δίκαιο με πολλούς τρόπους. Να πω όμως ότι αυτό δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τα σημεία 10 και 13 για την ε, Τουρκία τα οποία αντιβαίνουν στο άρθρο 47 του κανονισμού που λένε ότι το πρόεδρο, ε, του Κοινοβουλίου αποστέλει ένα θέμα ε, σε μια επιτροπή στις 4 Μαΐου Μαΐου υπήρξε μια ανακοίνωση που έλεγε ε, ότι κανένα θέμα δεν θα συζητηθεί σε επιτροπή αν δεν έχει σεβαστεί η Τουρκία τα 72 κριτήρια. Άρα μπορεί να γίνονται αυτά τα νομικά τεχνάσματα για να ε, σώσουμε την, ε, την συμφωνία, αλλά και η ίδια η ΛΥΜΠΕ παραβιάζει τον δικό μας κανονισμό με αυτό που κάνει. Αυτό έχει να κάνει και με το επόμενο θέμα, αλλά ε, θα ζητήσω από τον νομομαθή συνάδελφο πολύ σύντομα, μέσα σε 4-5 λεπτά, να σχολιάσει και καθώς το κάνει να μας επιβεβαιώσει ακριβώς τη φύση του θέματος ε, που εξετάζουμε σήμερα το βράδυ. Τι είναι σε επίπεδο νομικού καθεστώτος και πώς ε, πρέπει να το αστυνομεύσουμε, πώς να το αντιμετωπίσουμε εντός του νομικού συστήματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος και θα επανέλθω μετά από τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που έγιναν, καταρχάς, ε, στη νομική διάσταση αυτής της δήλωσης. Ε, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στο διεθνές ε, δίκαιο, διεθνή συμφωνία θεωρείται οποιαδήποτε δέσμευση λαμβάνεται μέσα στα πλαίσια ε, του ε, διεθνούς δικαίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. όποια διέσμευση λοιπόν αναλαμβάνεται από υποκείμενα του διεθνούς δικαίου που έχει μία δεσμευτική υποχρεωτική μορφή. Ε, όποια και αν είναι αυτή η δέσμευση, ε, όπως ε, είπαν και πολλοί από τους προηγούμενους που σχολίασαν, είμαστε σε μια φάση, λοιπόν, όχι μια ε, συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το νομικό ζών που εξετάζουμε σήμερα, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, δεν μας κάνει να μην το θεωρούμε διεθνή συμφωνία. Χρειάζονται βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να δούμε αν είναι διεθνή συμφωνία. Καταρχάς, η θέληση των μερών ε, απαιτείται. Που, η θέληση των μερών που υπέγραψαν τη συμφωνία. Το θέμα εδώ είναι αν θεωρούν τα μέρη ότι δεσμεύονται από αυτή τη συμφωνία σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και η πρόθεση των μερών έχει ως αποτέλεσμα ταυτόχρονα και τους όρους της συμφωνίας αλλά και τις συνθήκες ε, υπό τις οποίες ε, πέρασε αυτή η συμφωνία. Ε, αν δούμε λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη εξέταση, ε, είναι δύσκολο να καταλήξουμε εάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία θέλησαν νομικά να δεσμευτούν από αυτή τη δήλωση. Ε, το πρώτο στοιχείο που μας πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι η μορφή που επελέγει, ε, που ήταν η θελημένη από τα δύο ε, μέρη. Πρέπει να παρατηρήσουμε, να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η δήλωση ήταν απλώς μια ανακοίνωση τύπου που στην ουσία δεν έχει και καμία υπογραφή επάνω της. Αυτή η δήλωση δεν δημοσιεύθηκε πουθενά σε καμία επίσημη εφημερίδα. Ε, για παράδειγμα, στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στη δήλωση ε, δεν μας παραπέμπει καθόλου στα στάνταρ που νομικά χρησιμοποιούνται στις διεθνείς συμφωνίες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όμως πραγματικά μπορώ απέχει από τα πρότυπα σύνταξης μιας διεθνούς συμφωνίας. Ε, άρα από νομική άποψη δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι εδώ έχουμε μία διεθνή συμφωνία υπό την έννοια του άρθρου 218 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είχαμε κάτι τέτοιο, οι διαδικασίες ε, ε, δεν θα... Θα έπρεπε να είναι διαφορετικές. Δεν έχουμε όμως μια τέτοια συμφωνία. Τώρα ένα άλλο ζήτημα που θέλω να επαναλάβω μετά από τις παρατηρήσεις είναι ε, το τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο σε αυτό το στάδιο. Είπα ε, κατά την παρέμβασή μου ότι μετά από αυτή τη δήλωση ε, ακριβώς πρέπει να υιοθετηθούν κάποιες πράξεις μέσα από τις οποίες ε, το Κοινοβούλιο θα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Ανέφερα την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις θεωρήσεις. Αυτή η τροποποίηση πρέπει να γίνει μέσω της συναπόφασης. Άρα το Κοινοβούλιο στην ουσία θα πρέπει να δει αν τα 72 κριτήρια αναφοράς ε, που αναφέρονται στην ίδια τη δήλωση και η οποία δήλωση λέει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά για να μπορέσουμε να άρουμε τις υποχρεώσεις για τις θεωρήσεις. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να εξετάσει αν αυτά τα 72 κριτήρια γίνονται σεβαστά και αν καταλήξει ότι δεν γίνονται σεμβαστά, πρέπει αντίστοιχα να ψηφίσει. Ε, το Κοινοβούλιο επίσης πρέπει να γνωμοδοτήσει μέσα στα πλαίσια της απόφασης που έχει λάβει το Συμβούλιο για την ε, επανακατανομή των προσφύγων, ε, την επανεγκατάσταση δηλαδή, που με την κατάσταση των προσφύγων. Έτσι μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας ε, του προϋπολογισμού θα πρέπει να αποφασίσει και για την επανακατανομή των πόρων που ε, σχετίζονται με το θέμα αυτό όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει πολύ πολύ σύντομα να αναφέρω πριν ολοκληρώσω είναι κατά πόσο αυτή η δήλωση συνάδει με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, αν συμπορφώνεται με το δίκαιο αυτό. Το ζήτημα αυτό ε, δεν τίθεται όταν μιλάμε για πραγματική συμφωνία. Όμως αυτή η δήλωση δεν είναι μια ε, νομικά δεσμευτική πράξη, δεν είναι συμφωνία. Οπότε δεν, ε, αλλιώς, γι' αυτό το λόγο σκεφτόμαστε γιατί αν σέβεται ή όχι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είπα λοιπόν στην πρώτη μου παρέμβαση ότι αυτή η δήλωση δεν έχει σκοπό να τροποποιήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και συγκεκριμένα μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για την επιστροφή, η οποία δεν τροποποιείται με αυτή τη δήλωση. Άρα οι υποχρεώσεις που ε, προβλέπει αυτή η οδηγία συνεχίζουν να ισχύουν και στη φάση της εφαρμογής των μέτρων που αναφέρει η δήλωση θα πρέπει κανείς να ε, διαπιστώσει εάν όντως ε, αυτές οι, αυτά τα μέτρα εσέβονται τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Ευχαριστώ. Με ενθαρρύνει με το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε πολύ νομική δουλειά να κάνετε εσείς και οι συναδελφοί σας και το λέω αυτό ως ε, ε δικηγόρος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο Concord, όχι αεροπλάνο, το παλιό αεροπλάνο, αλλά μια σύμπνια, αν θέλετε. Σίγουρα θα έχουμε και άλλα σχόλια. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας πάντα. Προχωρούμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο θέμα μας. Την περασμένη εβδομάδα πήραμε από την Επιτροπή ένα πακέτο εγγράφων για την απελευθέρωση των θεωρήσεων που προανέφερα ε, ως προς την Τουρκία που περιλαμβάνουν την τρίτη έκθεση πρόεδρου, πρόδου, το έγγραφο εργασία, πρόταση τροποποίηση του κανονισμού 539 του 2001 για την Τουρκία και μια επιπλέον πρόταση τροποποίηση του κανονισμού 539 για την τροποποίηση του υφιστάμενου μηχανισμού αναστολή. Το θέμα συζητήθηκε και στη διάσκεψη των Προέδρων που από πλευρά του επέμεινε να τηρηθούν όλα τα ορόσημα από την Τουρκία μέχρι ότου συμβεί πλήρω κάτι τέτοιο και μέχρι ότου η Επιτροπή παράσχει στο Κοινοβούλιο γραπτή εγγύηση ότι τούτο συμβαίνει. Θα πρέπει να συνεχιστεί η πλήρης ε, ε, ε, ενασχόληση με το θέμα αυτό χωρίς παραπομπή σε επιτροπή. Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα τις εργασίες μας και δώσω το λόγο στην κυρία Τσίγκαν για μια παρουσίαση των διαφόρων κειμένων κατόπιν μέσα στο όριο του χρόνου μας θα επιτρέψω στα μέλη που θέλουν να λάβουν το λόγο να το κάνουν. Η κυρία Τσιγκάν λοιπόν έχει πρώτα το λόγο. Το λόγο για μια σύντομη σχετικά αλλά σημαντική παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Γεια σας αγαπητά μέλη της Επιτροπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να παρουσιάσω την έκθεση και την νομοθετική πρόταση για την Τουρκία για την απελευθέρωση της βίζας ε, που υιοθέτησε η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπατε. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια σύντομη εισαγωγή των ε, κειμένων αυτών που μόλις εγκρίθηκαν από το Σώμα των Επιτρόπων. Το πρώτο και δεύτερο έγγραφο αφορά την τρίτη έκθεση που αξιολογεί την πρόοδο της ε, Τουρκίας ε, όσον αφορά τα 72 κριτήρια του οδικού χάρτη του Δεκεμβρίου 2013. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από ένα έγγραφο εργασία της ε, Κομισιόν που δίνει λεπτομερείς εξηγήσει για το κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια. Τα δύο αυτά έγγραφα, η έκθεση και το έγγραφο εργασίας ε, πηγαίνουν μαζί. Και έτσι πρέπει να τα δείτε. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει στην Επιτροπή και είχα την ευκαιρία και την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω τη δεύτερη έκθεση, συζητήσατε την ε, δεύτερη έκθεση που αφορούσε την κατάσταση αρχές Μαρτίου φέτος. Εν τω μεταξύ, πέρασαν δύο μήνες, η απαλλαγή από βίζα, όπως συζητήσατε, ε, έγινε ένα βασικό στοιχείο μετά την ε, συνάντηση της 18ης Παρτίου και τέθη μια προθεσμία η οποία είναι το τέλος Ιουνίου για να ολοκληρωθεί ο δικός χάρτης. Στην διαδικασία λοιπόν αυτή η απελευθέρωση της βίζας ε, έχουν αναλυφθεί πολλές μεταρρυθμίσεις από τις τουρκικές αρχές και είτε συνεχίστηκαν είτε ξεκίνησαν ε, νέες και αυτά είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην επιτάχυνση της υιοθέτησης των σχετικών μέτρων. Στην τρίτη έκθεση η Κομισιόν αναφέρει τα αποτελέσματα αυτής της επιτάχυνσης και τα αποτελέσματα είναι υποσχόμενα. Η Τουρκία μέσω των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων ή και των νέων μεταρρυθμίσεων έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο και όλοι ξέρουμε πως η διαδικασία αυτή είναι ένα στέρεο πλαίσιο που μας βοηθάει να επιτύχουμε μεταρρυθμίσεις σημαντικές για τους πολίτες και τις οικονομίες ε, και των δύο πλευρών. Είναι ένα σημαντικό μέσο το οποίο μας επιτρέπει στα πολιτικά δηλαδή και νομικά συστήματα να προσεγγίσουν με τις προδιαγραφές της Ένωσης και είναι ακριβώς αποτελεσματική και οι μεταρρυθμίσεις είναι μόνιμες. Σε προηγούμενη συνεδρία, όταν συζητήσαμε την δεύτερη έκθεση αναφέρθηκα στα κεφάλαια της απελευθέρωσης βίζας ε, και της σχετικής έκθεσης πρόοδου Προσπάθησα να σας δώσω κάποια θετικά παραδείγματα των όσων έχουν ήδη γίνει και ανέφερα και κάποια στοιχεία τα οποία προφανώς έπρεπε να εκπληρώσει η Τουρκία σήμερα. Θα κινηθώ αλλιώ να αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην έκθεση και μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή στο έγγραφο εργασίας. Θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα των θετικών εξελίξεων και μετά θα εστιάσω σε 7 συγκεκριμένα κριτήρια. Παραδείγματα των επιτευγμάτων των θετικών των τουρκικών αρχών. Ενίσχυσαν την ποιότητα των δελτίων ταυτότητας και άρχισαν να μοιράζονται πληροφορίες με τα κράτη-μέλη για τα πλαστά έγγραφα. Επίσης συνεργάζονται πλήρως με την Ελλάδα όσον αφορά τη Συμφωνία Επανεισδοχής και έχουν μειώσει τον αριθμό αφήξεων στην Ελλάδα από 6.000 την ημέρα τον Οκτώβριο 2015 σε 140 τον Απρίλιο φέτος. Φιλοξενούν ε, γύρω στα 3 εκατομμύρια πρόσφυγες ε, με πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση και σε νόμιμη απασχόληση και μειώνουν σταδιακά την καθυστέρηση που υπάρχει στην επεξεργασία των αιτήσεων σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα. Έχουν κυρώσει τις ε, συμβάσεις Συμβουλίου της Ευρώπης και τα πρωτόκολλα της Χάγης και ενέκριναν ένα νέο νόμο περί διακίνησης ανθρώπων ε, και επίσης ενέκριναν σχέδια δράσης για τα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα, την διαφθορά και την παράτυπη ανάσταση. Και αυτά είναι κάποια παραδείγματα για να δούμε όλα αυτά. Κριτήρια, βεβαίως, ε, για να τα δείτε αυτά πρέπει να ανατρέξετε στο έγγραφο εργασίας για να τα δείτε λεπτομερώς. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε κάποια κριτήρια τα οποία είναι ιδιαίτερα γιατί αντικειμενικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για εφαρμογή για διάφορους λόγους, πρακτικούς και διαδικαστικούς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στην αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομετρικών διαβατηρίων που περιλαμβάνουν κάποια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία θα αρχίσει να τα εκδίδει τον Ιούνιο. Ακόμα λοιπόν και αν χορηγηθεί ε, καθεστώς ε, τέτοιο ε, απαλλαγής από τη Βίζα στη ε, Τουρκία μόνο οι κάτοχοι των νέων διαβατηρίων θα μπορούν να μπουν στην ζώνη Σέγγεν χωρίς Βίζα. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο ήθελα να αναφέρω αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας Πανεσδοχής που θα συμπεριλαμβάνουν και την επανεισδοχή υπηκών τρίτων χωρών. Γνωρίζουμε όλοι ότι αρχικά οι διατάξεις για τους υπηκούς τρίτων χωρών θα έπρεπε να έχουν τεθεί ενισχύ σε ένα χρόνο το καλοκαίρι του 2017. Οι τουρκικές αρχές έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις για την επανεισδοχή υπηκών τους από τον Οκτώβριο του 2014 αλλά για τους υπηκόους τρίτων χωρών επιτάχυναν την ημερομηνία 1η Ιουνίου 2016, αλλά προφανώς η θέση ενισχύ ενισχύει ειναι την 1η Ιουνίου, οπότε σημαίνει πως τον Ιούνιο θα δούμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε πέντε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία σαφώς δεν εκπληρώνονται και τα οποία περιγράφουμε στην έκθεση και στο έγγραφο εργασία. Αφορούν πρώτα απ' όλα τα μέτρα τα οποία αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πρόληψή της. Εδώ πέρα μιλάμε για αποτελεσματική συνέχεια των συστάσεων της ομάδας της Χάγης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το δεύτερο αφορά την προστασία δεδομένων και την ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσίας με την κοινοτική έτσι ώστε πρώτα απ' όλα ότι θα υπάρχει μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων η οποία θα είναι ανεξάρτητη και οι δραστηριότητες ε, των διοκτικών αρχών θα είναι εντός των πλαισίων του νόμου. Η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων επίσης επηρεάζει το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω που είναι η σύναψη μιας επιχειρησιακής συμφωνίας με την Europol. Οι διαπραγματεύσεις για την συμφωνία αυτή μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά την υιοθέτηση των απαραίτητων στοιχείων για την ομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το τέταρτο στοιχείο αφορά την αποτελεσματική δικαστική συνεργασία για ποινικά ζητήματα και τέλος η τρομοκρατία. Εδώ πέρα αναφέρομαι στην αναθεώρηση και της νομοθεσίας αλλά και της πράξης ε, για να ευθυγραμμιστούν αυτά με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το επίπεδο εμπλοκής λοιπόν και αποφασιστικότητας της ε, Τουρκίας νομίζω πως είναι απτό εάν δείτε την έκθεση και το έγγραφο εργασία. Βλέπετε διαφορά από τη δεύτερη έκθεση ε, πρόοδου και θεωρώ πως ε, εγκρίνοντας την έκθεση η Κομισιόν αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία για να ε, επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα και στα υπόλοιπα κριτήρια. Και ακριβώς η εκπλήρωση των υπόλοιπων κριτηρίων είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τα επόμενα βήματα όσον αφορά την έγκριση των σχετικών ε, νομοθετικών προτάσεων που επίσης είναι επιτάπητο σήμερα. Γνωρίζετε επίσης πως η Κομισιόν ταυτόχρονα παρουσίασε την πρόταση για να αλλάξει ο κανονισμός 539 για να φύ, πάει η Τουρκία στον κατάλογο χωρών που απαλλάσσονται από βίζα. Παρακολουθώντας τη συζήτηση σας πριν στο, για το σημείο 5 για την δήλωση της 18ης Μαρτίου το σημείο το οποίο αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης γίνεται αναφορά και στην σχετική απόφαση για την αλλαγή του κανονισμού. Υπάρχει μία σαφής αναφορά και παραπομπή στην διαδικασία που απαιτείται για να αλλάξει ο κανονισμός και παραπομπή στον ρόλο των συνομαστών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που όντως θα λάβουν την απόφαση. Οπότε η Κομισιόν ενέκρινε αυτή την πρόταση για να σεβαστεί την προθεσμία των 8 εβδομάδων για τη διαβούλευση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και για το λόγο αυτό έπρεπε η πρότασή μας να γίνει τώρα μαζί με την έκθεση η οποία περιέχει μια ακριβή και ειλικρινή περιγραφή της κατάστασης και συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι ε, σχεδιάζουμε να κάνουμε με τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες απαιτήσει. Γνωρίζουμε το ότι έχουμε πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα αλλά είναι σαφές ότι το σημείο αναφοράς για όλους μας είναι η ισχυρή βούληση να περιορίσουμε την χειρότερη μεταναστευτική κρίση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν πως σας παρουσιάζουμε ένα έγγραφο το οποίο έγγραφα, τα οποία είναι πολύ καλά προετοιμασμένα με βάση τις πληροφορίες που είχαμε και είχαμε μια ξεκάθαρη περιγραφή της κατάστασης. Ελπίζουμε να επιδείξει πνεύμα συνεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αναγκαία πολιτική βούληση ε, όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, ε, ο πρόεδρος, σας παρακαλώ, συντομεύετε, γιατί ε, έχουν μείνει μόλις 15 λεπτά για να μιλήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Για κάντε λίγο πιο γρήγορα λοιπόν. <clears throat> Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με τον τεινόμενο μηχανισμό αναστολής. Το τελευταίο νομοθετικό κείμενο δεν αφορά την Τουρκία. Τονίζω ότι αφορά οριζόντια όλες τις χώρες τις οποίες υπάρχει απελευθέρωση θεωρήσεων. Είναι, προβλέπεται ήδη στον 539. Η βασική στόχη της πρώτας επιτροπής στο θέμα αυτό είναι η εξής επιτάχυνση της διαδικασίας, μειώνοντας την περίοδο αναφοράς που προβλέπει ε, η διαδικασία σε δύο μήνες και προθεσμοί για την Επιτροπή για να υποβάλει την, την, ε, την εκτελεστική πράξη από τρει μήνες στον ένα μήνα για την υλοποίηση του μηχανισμού. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής ε, και των λόγων της αναστολής για να βελτιωθούν οι απορρίψεις ε, εισόδων από τρίτες χώρες και δίνει την δυνατότητα στην Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πέραν των κρατών μελών που ήδη είχαν τη δυνατότητα αυτή. Ακόμα και σε περίπτωση που μια τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται σε θέματα επανειδοχής. Με αυτά κλείνω την παρουσίαση και των τεσσάρων κειμένων Περιμένω σχόλια και ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε 16-17 λεπτά και 16-17 ομιλητές. Δεν θα πρέπει να ενημερώσω για τον Κλοντ και να του πω ότι δεν κατέληξε σε χάος. Αν κρατήσετε ένα-ενάμιση λεπτό ο καθένας, θα καλύψετε, θα μπορούσαμε να σας καλύψουμε. Αλλιώ θα σας κόψω. Συντονιστές θα μιλήσουν, αλλά θα το κάνω, παρότι θα γκρινιάσουν κάποιοι ξανά, εάν κρατήσουν τον χρόνο τους. Αλλιώ δεν θα αφήσουν τους άλλους να μιλήσουν και θα πρέπει να γκρινιάξουν στον συντονιστή τους. Η κυρία Χόλμαγερ πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι προσπαθούν ε, να ενισχύσουν τη συνεργασία με την Τουρκία και να μας πούνε ότι έχουν γίνει κάποιες προέδροι οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα που παραμένουν. Για παράδειγμα το θέμα της αντιπρομοκρατικής ε, νομοθεσίας, ειδικά ε, ως προς τους Κούρδους και τη μειονότητα των Κούρδων που χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο μηχανισμός μηχανισμός αξιολόγησης που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό είναι μια ε, θετική εξέλιξη ε, όσον αφορά στην απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αν θέλουμε να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε ε, τήρηση και των γεγονότων που έχουν να κάνουν τη συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουμε πρόσφυγες από την Τουρκία. Θα ήθελα να δω αν μπορούμε να ε, επιταχύνουμε τη διαδικασία επιλογής, να έχουμε δηλαδή νόμιμους ε, δρόμους για να μπορούν οι άνθρωποι να έρχονται σε εμά έτσι και να μην ε, υπάρχουν κίνητρα για τους παράνομους μετανάστες. Να υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία. Πώς έχουμε προχωρήσει ως προς αυτή την νόμιμη οδό ε, για τους ε, ε, πρόσφυγες. Όπως είπε και η συνάδελφος Άννα Γκόμες, θα, έπρεπε, θα μπορούμε να πάρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ο καθένας στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σίπελ, έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος, όμως μάλλον στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Αυτό Φαίνεται ότι αυτοί που έχουν βιομετρικό διαβατήριο μόνο μπορούν να ε, ταξιδεύουν χωρίς βίζα. Είμαστε σίγουροι ότι η Τουρκία θα δίνει σε όλους τους πολίτες της τέτοια διαβατήρια ή μόνο σε αυτούς που τις αρέσουν. Θα ήθελα περισσότερη πρόοδο στην πράξη και όχι στα χαρτιά. Το ίδιο και για τον αντιπροτρομοκρατικό νόμο. Φαίνεται ότι δεν, είναι, δεν προτίθεται να αλλάξουν τίποτα. Ε, τώρα, για την προστασία των δεδομένων για την ανεξαρτησία. Ακόμα και το νομικό και το αστυνομικό σύστημα στην Τουρκία ε, δεν είναι ανεξάρτητο. Γιατί να είναι η αρχή προστασίας δεδομένων ανεξάρτητη λοιπόν δεν έχουμε ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της έκφρασης. Είδατε τι συνέβη σε κάποιους δημοσιογράφους που απλώς ανέφεραν γεγονότα. Τώρα ρισκάρουν να μπουν στη φυλακή για πέντε χρόνια ή περισσότερο. Και για τον μηχανισμό Ε, είναι πολύ καλός από όσο έχω διαβάσει, όμως τον σκεφτόμαστε ε, μόνο όταν πολλοί μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη από αυτή τη χώρα. Δεν μιλάμε για θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και αν γίνονται σεβαστά. Ε, άρα πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα και δεν έχω πιστεί ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι όσον αφορά εμά και τη δική μου ομάδα, το... οποιαδήποτε πρόοδος ως προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων προς την Τουρκία θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των κριτηρίων. Ε, το να είμαστε κοντά ή να λέμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα ε, πληρούνται ε, δεν αρκεί. Πρέπει να έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω, αλλά να μην δίνουμε τέτοιες ανταμοιβέ. Κάτι ε, τέτοιο θα στείλει λάθος μήνυμα σε πολλές άλλες χώρες που μπορεί να θεωρούν ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση προς την Τουρκία και ότι τους ε, βλέπει διακριτικά. Τώρα, αυτό ήθελα να πω η κυρία Βίλστρομ, ε, λίγο σύντομα. Ευχαριστώ, Τίμωθη. Συμφωνώ πλήρως με πολλά από αυτά που μόλις ανέφερες. Όταν έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια, τότε θα μιλήσουμε, όχι πριν από αυτό. Επίσης, εκπλήσωμαι από το γεγονός ότι η έκθεση πρόοδου δεν περιλαμβάνει ούτε μία λέξη για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, παρόλο που μιλά για νομοθετικά ε, μέτρα κανείς αναρωτιέται αν η Κομισιόν δεν έχει δει καν ότι υπάρχει αύξηση στην καταστολή των μειονοτήτων, των ακαδημαϊκών, των blogger και οποιοδήποτε πνευματικών ανθρώπων είναι αντίθετη με ε, τον, κύριο Ερντογάν. Η Κομισιόν καταλήγει ε, λέγοντας κάτι που είναι πραγματικά ε, ανήκουστο. Λέει ότι χρειάζεται περισσότερη ε, πρόοδος για κάποιες εξαιρετικές απαιτήσει που, απομένουν. Ε, είναι τραγωδία αυτό. Όσον αφορά για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ε, δεν υπάρχει ούτε καν αναφορά ε, το πυροβολισμού δηλαδή, που σκοτώνουν τους πρόσφυγες ε, στα σύνορα της Τουρκίας δεν αναφέρει ε, ξεκάθαρα ότι η Τουρκία δεν έχει σκοπό να εκπληρώσει τα κριτήρια, λέει απλώς ότι δεν τα έχει εκπληρώσει. Πώς ε, δίνουν λοιπόν αυτή την πρόταση για να έχουμε άρση των θεωρήσεων το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει αυτό το βήμα ε, ε, και να εμπιστευτεί την Κομισιόν. Ε, πώς να την εμπιστευτούμε ότι δεν θα κάνει και άλλες τέτοιες συμφωνίες, τέτοια κατασκευάσματα με την Τουρκία. Μόλις εκπληρώσουν λοιπόν οι Τούρκοι τα κριτήρια, με μεγάλη μας χαρά να απελευθερώσουμε τις θεωρήσεις. Αλλά όχι πριν από αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ένστ. Όχι, Σπινέλη. Ευχαριστώ. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν την περασμένη Παρασκευή ανέφερε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει την νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας. Θα συνεχίσουν να θεωρούνται δηλαδή ως τρομοκράτες οι δημοσιογράφοι, οι αντιφρονούντες, οι Κούρδοι αγωνιστές, οι πανεπιστημιακοί που επικρίνουν την κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω την κυρία Τσιγκάν της Επιτροπής είναι μπορεί να διευκρινίσει τι συμβαίνει αν σημαντικά benchmark, ορόσημα, κριτήρια για την απελευθέρωση των θεωρήσεων δεν ε, τηρηθούν. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κριτήρια. Κάτι ακόμα. Θα ήθελα από σεβασμό προς το Κοινοβούλιο να μας πει ξεκάθαρα και με διάφανο τρόπο πώς τηρούνται και τα 72 benchmark. Γίνονται σεβαστά. Ξεκάθαρα. Γιατί τα λόγια της Επιτροπής για την Τουρκία αφήνουν πολλά κενά. Σας θυμίζω ότι ο Τίμερμαντς είπε ότι η πρόοδος ε, που έχει επιτύχει η Τουρκία είναι θεαματική, θεαματική. Θυμίζω για την αντιμετώπιση των προσφύγων μία προφράση του Ντόναλτ Τούσκ από τις 20 Απριλίου. Η Τουρκία, και παραθέτω, είναι το καλύτερο παράδειγμα στον κόσμο για το πώς αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες. Το καλύτερο παράδειγμα στον κόσμο. Ρωτώ την Επιτροπή να μας εξηγήσει αυτά τα 72 benchmark και να δει την πραγματικότητα μιλώντας για το τι πραγματικά γίνεται στην Τουρκία. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό θα έχει η Κομισιόν, οπότε πολύ δύσκολα θα μπορεί να εξηγήσει και τα 72. Η κυρία Βαλέρο για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ως πράσινη είμαι γενικά υπέρ της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Δύσκολο μπορώ να το κάνω αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η συμφωνία με την Τουρκία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι δύσκολο να μιλήσω λοιπόν επενώντας την ε, απελευθέρωση. Θα ήθελα να δω το κριτήριο υπαριθμών 65 που αναφέρει η Κομισιόν το λέει ότι δεν τηρείται το κριτήριο. Σε κάποια λέει εν μέρη τηρούνται, εν μέρη υλοποιήθηκαν, ε, σχεδόν υλοποιήθηκαν. Αυτό το κριτήριο το 65 δεν τηρείται. Πώς θα υλοποιήσει η Επιτροπή Πώ θα φροντίσει η Επιτροπή να υλοποιήσει η Τουρκία αυτό το κριτήριο, ιδίω με δεδομένο ότι ο Έντογκαν είπε ότι δεν έχει στόχο να αλλάξει την νομοθεσία για την δημοκρατία που είναι το θέμα, το αντικείμενο του κριτήριου 65. Ευχαριστώ. Η κυρία Ο κύριο Λεμπρετών, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα 72 κριτήρια επί ούτε πρόκειται να το κάνει. Η Ένωση θα συνάψει λοιπόν μία συμφωνία παραβιάζοντας τις αξίες και το νομικό της πλαίσιο. Για την διαδικασία είναι εντυπωσιακό το ότι μιλάμε για το θέμα αυτό. Επανέρχομαι στην, στον ανακοινωθέν της 4ης Μαΐου που λέει η διάσκεψη των Προέδρων δεν θα υπάρξει επιστροφή στις επιτροπές ενώσο δεν πληρούνται τα 72 κριτήρια διηνθάτερον ή παραβιάζουμε ρητά και εσκεμένα τις ε, ε αποφάσεις της διασκεψης των Προέδρων ή και αυτό είναι που θεωρώ πιο πιθανό ακούγοντα την απάντησή σα, Πρόεδρε, είναι ότι η ανακοίνωση αυτή είναι μια παγίδα, ένα ψέμα για να εξαπατηθεί η κοινή γνώμη τη Ευρώπη. Η τελευταία φράση που αναφέρω δεν, μπορεί, δεν μπορεί να υπάρξει καμία αναπομπή σε επιτροπή, αντί ε, αντιβαίνει στην προηγούμενη που λέει θα πρέπει να συνεχιστούν οι ε, διεξοδικές διαπραγματεύσεις. Ο τύπος θα νομίσει ότι πρόκειται για διαπραγματεύσεις ενώ εσείς λέτε ότι η Επιτροπή μπορεί να δράσει. Αυτό είναι επέσχυντο. Δεν θα πείσετε τη γαλλική τουλάχιστον κοινή γνώμη. Εγώ ξεκαθάρισα ότι μπορεί να συνεχιστεί η περαιτέρω δουλειά αλλά δεν θα υπάρχει αναπομπή σε επιτροπές. Το είπα. Έχουμε τέσσερα λεπτά πέντε άτομα και απάντηση επιτροπής. Ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να θυμίσω σε ε, συναδέλφους ότι δεν ξέρω τα γεγονότα με Σίλια Μάνστρομ έχει ε, υπογράψει το Δεκέμβριο του 2013 μια συμφωνία με την Τουρκία. Ήταν η συμφωνία επανεσδοχής έναντι της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Αυτή η διαδικασία ήταν η πιο αργή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επανήλθε τώρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο δράσης με... στην Τουρκία διότι ε, είχαν παγώσει αυτές οι διαδικασίες που δεν έχει συμβεί με κανένα άλλο κράτος. Η ε, θεώρηση, η, απελευθέρωση των θεωρήσεων έχει να κάνει με την επαφή μεταξύ ανθρώπων. Ήμουνα σκιώδης εισηγήτρια για την Βοσνία και όλη η Ενωμένη Αριστερά έλεγε από την ε, λευκή λίστα, από την, στη μαύρη λίστα για να ξεχάσουμε το Σαράγεβο τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να κάνουμε ένα, μια πολιτική κίνηση. Όμως εγώ έλεγα ότι πρέπει να τηρούμε τα κριτήρια και τον οδικό χάρτη, να σταματήσουμε την επιθετικότητα, τον θυμό και την τιμωρητική στάση, γιατί τιμωρούμε τον κόσμο και όχι τον Ερδογκάν θα πρέπει να, ε, μάλλον να ξεχνάμε ότι έχουμε δώσει ε, απελευθέρωση σε 55 χώρες όπως την απόλυτη ε, μοναρχία του Βρουνέη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και άλλες τέτοιες χώρες που δεν έχουν λιγότερες, λιγότερα προβλήματα. Δεν πρέπει να έχουμε πιο αυστηρά στάνταρ για την Τουρκία. Ο κύριος Νταβούτογλου, αυτός παρετήθηκε ε, γιατί αυτός ε, ε, αναγκάστηκε να το κάνει επειδή εμείς έχουμε αυτή τη στάση στο Κοινοβούλιο υποσκάπτουμε τους ε, μετριοπαθείς στην Τουρκία. Ο κύριος Λένος, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι ως τώρα ε, μίλησαν για τα 72 κριτήρια που πρέπει να πληρούνται πριν να ξεκινήσουν συζητήσει για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Όμως Πότε βλέπουμε ότι τηρείται ένα κριτήριο, ας πούμε, ε, όταν έχουμε τα βιομετρικά διαβατήρια ή την αντιτρομοκρατική διαδικασία, ε, νομοθεσία ή την νομοθεσία κατά των διακρίσεων, απλώς ε, βάζουμε ένα σταυρό σε ένα κουτάκι. Είναι δύσκολο. Σε αυτό το κοινοβούλιο τα τελευταία έξι χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με Τούρκους υπουργούς για αυτά τα τρία νομοθετικά ε, ζητήματα και μας εξήγησαν πολλές φορές γιατί ήταν δύσκολο ή αδύνατο να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στην Τουρκία. Και τώρα μέσα σε τρεις εβδομάδες θα καταφέρουν να ε, εγκρίνουν νομοθεσία που θα πάει τόσο μακριά και θα αγγίζει τα θεμελιώδη προβλήματα στην Τουρκία. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω και δεν ξέρω ε, πώς το Κοινοβούλιο θα ελέγξει όχι μόνο τα χαρτιά, αλλά την πράξη να δούμε τι σημαίνει όταν τικάρουμε ένα κουτάκι. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ζητώ συγγνώμη για τους υπόλοιπους ομιλητές που δεν θα μιλήσουν. Μόνο δύο-τρία μέλη θα μιλήσουν τώρα. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τσίζεκ. Uh, θα σας διευκολύνω, δεν ζήτησα το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν για την προηγούμενη συζήτηση. Ορίστε λοιπόν. Ε, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαυρίδης τώρα. Σας ε, ε, υποσχέθηκα να πείτε κάτι. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Επίσης, αν κάποιος αισθάνεται ένοχος για το συμβαίνουν στην Τουρκία ή για τον Ερντογάν, είναι δικό του πρόβλημα, η δικό της. Εμείς εδώ πέρα πρέπει να υπερευθυστούμε τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την αξιολόγηση της Κομισιόν. Ε, θα αναφερθώ σε ένα κριτήριο μόνο. Ένα από αυτά που έχει μάλιστα εκπληρωθεί κιόλα. Το υπαριθμόν 44. Με βάση την αξιολόγηση έχει εκπληρωθεί. Και τέλος τέλος, στην παράγραφο, στο κάτω κάτω μέρος, λέει πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η Τουρκία δεν συνεργάζεται καθόλου με την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της πολιτικής της ε, μη αναγνώρισης. Μπορώ να σας πω και άλλα. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Είμαστε 28 ισότιμα κράτη-μέλη ή όχι. Πιστεύουμε στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σοφή Ινετφέλτ για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα πως εγώ ήμουν πάντα υπέρ της απολευθέρωσης βίζας με Τουρκία αλλά η διαδικασία έχει γίνει πλέον ε, πολύ περίεργη. Η κυρία Κόρτσαπέλτ είπε πως δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν ε, να κάνουμε ε, για την Τουρκία ότι κάνουμε και για τις άλλες χώρες. Υπάρχουν 72 κριτήρια, πρέπει να εκπληρωθούν. Απλό είναι. Και τώρα η Κομισιόν μας λέει πως ε, δεδομένη στις ευαίσθητες φύσης ε, του θέματος θα έπρεπε να έχει έρθει εδώ πέρα ο ίδιος ο Επίτροπος αντί για κάποιον υπάλληλο. Ε, τέλος η Κομισιόν λέει ότι έχουμε πιεσμένο χρονοδιάγραμμα. Ε, με συγχωρείτε, το χρονοδιάγραμμα δεν είναι πιεσμένο ε, λόγω της διαδικασίας αυτής, αλλά επειδή η Κομισιόν το συνέδεσε με το προσφυγικό. Ενώ είναι δύο διακριτά ζητήματα. Οπότε, όπως λέει και η κυρία Κορατσαμπίλ, θα κάνουμε τη διαδικασία κανονικά και θα κρίνουμε το εάν η Τουρκία εκπληρώνει τα κριτήρια ή όχι. Αυτό και μόνο και όχι με βάση το προσφυγικό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κριστοφόρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα υποβάλω ένα ερώτημα προς όλους και ιδιαίτερα προς την Κομισιόν. Υπάρχει κανένας πραγματικά που πιστεύει ειλικρινά με τα κριτήρια που υπάρχουν κάτω, έστω και αν η Τουρκία φαίνεται ότι τυπικά τα εγκρίνει και τα περνά νομοθετικά, ότι θα τα υλοποιήσει στην πράξη. Το δεύτερο και σημαντικό. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιου μεγάλου βαθμού και τόσων τεράστιων συνεπειών, όταν μια χώρα όπως την Τουρκία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνείται να αποδεχθεί ότι υπάρχουν 28 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θα αρνηθεί να εφαρμόσει τη Συμφωνία Επανεισδοχή. Όταν αρνείται να συνεργαστεί με αυτή τη χώρα, που είναι και γειτονική και έχει σχέση και με το προσφύγο. Πώ είναι δυνατόν η Κομισιόν αλλά και τα νομικά συμβούλια να αποδέχονται την Τουρκία να τηρεί αυτή την αρνητική, την παράνομη στάση, την παράνομη για τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στάση και να υπογράφουν μαζί συμφωνίε υπέγραψαν και άλλε συμφωνίε με την Τουρκία και δεν τι υλοποίησαν. Απλώ θέλουμε να υποκρινόμαστε. Θέλουμε να μην καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία παρανομεί όταν δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η άρση των θεωρήσεων χωρί την αναγνώριση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να απαντηθεί επιτέλου. Ευχαριστώ Thank you. Mrs. Gomez, one minute, please. Thank you. Κυρία Γκόμες, ένα λεπτό. Η εντολή του Κοινοβουλίου είναι πολιτική αξιολόγηση, ανεξάρτητα από τα τεχνικά κριτήρια και το αν πληρούνται ή όχι. Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίσουμε το γεγονός ότι στο θέμα αυτό έγιναν μεγάλες ε, υποχωρήσεις στον τομέα της, ε, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν φταίει η Ευρώπη που έδιωξε τον ε, κύριο Νταβούτογλου εντογαν Το θέμα δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και η πολιτική διάσταση. Ο Τσαντούλντα, ο δημοσιογράφος που δικάζεται, δικάζεται γιατί εξέθεσε το γεγονός ότι η Τουρκία, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν συνεργαστεί ε, με το ISIS και άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν να αγνοήσουν τα κράτη-μέλη μας. Κύριε Τσίγκαν, τι να μας πείτε τώρα κι εσείς σε τρία λεπτά, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σχολιάστε ίσως. Ούτε στο νομοθετικό κομμάτι δεν πήγαμε ακόμα. Έχουμε πολλούς άλλες ευκαιρίες να το κάνουμε μαζί σας και τους αδέλφους σας, αλλά αν μπορείτε, σε δύο λεπτά μπορείτε να συνοψίσετε. Αν δεν μπορείτε, εντάξει, δεν πειράζει, χάθηκε ο κόσμος. Ευχαριστώ. Θα είμαι, θα είμαι σύντομη. Έχω παρουσιάσει την έκθεση πρόοδου και παλιότερα στην Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, το είπατε κι εσείς, η διαδικασία απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι μια ένα στέρεο πλαίσιο πρόοδου. Πρέπει να κοιτάμε λοιπόν το θέμα της πρόοδου. Μιλάμε για 72 ορόσημα. Αν δείτε προσεκτικά την έκθεση, το Staff Working Document, το τελευταίο που εκδώσαμε, που δεν είναι σύντομο, περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση, έντιμη Μιλήσατε για την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Είναι στις τελευταίες σελίδες της έκθεσης, όπου λέμε η Επιτροπή καλύπτει τις ειδικές αρχές να προχωρήσουν μετά τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής τα μέτρα που είναι αναγκαία για να υλοποιήσουν τα εκρεμή ορόσημα. Αυτό αφορά την δημοκρατία. Αλλά έχει γίνει πολλή δουλειά. 72 ορόσημα είναι. Έχουν, έχουν ε, επικυρωθεί συμβάσεις. Έχουν τεθεί τα εργαλεία της, της ε, Έχετε το θέμα της υλοποίησης όντως, αλλά η νομοθεσία υιοθετείται. Έχουμε εξετάσει κάποιους από τους νόμους. Κάποια νομοθετικά κείμενα για την προστασία δεδομένων δεν τηρούν πλήρως τις υποχρεώσεις, αλλά ναι. Έχουμε συνεργαστεί με τους ομόλογους μας στην Επιτροπή για το backlog και θα δείτε ότι στο συγκεκριμένο ορόσημο περιγράφεται η δουλειά που γίνεται και τα αποτελέσματα. Ε, έχουμε πολλά θετικά ε, στοιχεία πρόοδου που πρέπει να τα δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων με την Τουρκία και την ε, επίλυση των κρίσεων, της κρίσεως. Εάν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και τα δούμε προσεκτικά και σας εξηγήσω και το πλαίσιο για μια σειρά ε, επικρίσεων, ερωτημάτων, σχολείων που έχετε, θα σας διευκολύνω και τη δική σας ανάγνωση. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας πείσουμε περισσότερο για τη δουλειά που γίνεται, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε και μια πιο θετική ατμόσφαιρα για το έργο αυτό, γιατί είναι μια πρόοδος που συμβαίνει στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, για τα οποία η μεθοδολογία δεν άλλαξε, θα συνεχίσει να παρακολουθείτε στην Επιτροπή. Νομίζω ότι θα μπορούσα να καλύψω και άλλα θέματα, αλλά δεν μου δώσετε πολύ χρόνο. Αυτή είναι η δική μου σύνοψη και συνιστά ταυτόχρονα και μια πρόσκληση να έθετε, θέλετε, να συζητήσουμε με βουλευτές ομάδες για τα διάφορα αυτά θέματα. Δείτε και την τελευταία, το τελευταίο τμήμα της έκθεσης, τα συμπεράσματα. Εκεί υπάρχουν σαφή σενάρια για μας, μια έντιμη παρουσίαση των επόμενων βημάτων. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για απευθείας συζητήσεις αν ε, θέλετε να δούμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι η δουλειά συνεχίζεται. Ο χρόνος περνάει. Ευχαριστώ. Επόμενη συνάντηση κυρίες και κύριοι, 23 Μαΐου. Δευτέρα, 3 με 6,5 και Τρίτη 9 με 12,5. Ευχαριστώ. Πέρας της συνεδρίασης.